Τώρα περνάμε στην δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Connecting Europe μετά από το 2020. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Μπολτ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας όσον αφορά τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη μετά το 2020. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο κανονισμό ε, περιλαμβάνεται και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε ήδη στις 2 Μαΐου που αναφέρει και τις προτεραιότητες του σχεδίου αυτού. Όλοι έχουμε υπόψη μας πόσο πολλές επενδύσεις χρειάζονται για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Για την περίοδο λοιπόν 2021-2027 πιστεύουμε ότι το, η ανάπτυξη του δικτύου αυτού θα χρειαστεί 350 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Επιπλέον πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο αποφασιστικά και την πρόκληση λιγότερος άνθρακας έως καθόλου άνθρακα στις μεταφορές αποτελεί βασικό στοιχείο του τι θέλουμε να καταφέρουμε. Επίσης, η κινητικότητα πρέπει να είναι ευφυής, βιώσιμη, για όλους, ασφαλής και γι' αυτό ακριβώς πρότεινα να εξυγχρονίσουμε τη διευκόλυνση αυτή ιδέα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα από τα λίγα προγράμματα για τα οποία έχει προταθεί αύξηση στον προπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για 42,3 δισεκατομμύρια, από τα οποία 30,6 θα πάνε στις μεταφορές. Η πρότασή μας ε, λοιπόν είναι να διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα προπολογισμού και για το γενικό φάκελο και για την συνοχή. 11,3 για τη συνοχή. Για παράδειγμα, επιπλέον θέλουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε για υποδομές μεταφορών διπλής χρήσης και στρατιωτικής και μη στρατιωτικής. Εδώ τώρα θέλω να αναφερθώ στα ποσά που αναφέρει το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις προτεραιότητες, συμφωνώ απόλυτα για το ότι είναι σημαντικό να έχουμε την καλή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη νέων υποδομών και τον εξυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων υποδομών. Από τη μια, συμφωνώ ότι πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του δικτύου για να καλυφθούν τα κενά. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί συνέχεια για να πετύχουμε τα μεγάλα σχέδια που προβλέπονται στο σημερινό πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη σημασία στον εξυγχρονισμό των υποδομών που ήδη υπάρχουν. Πρέπει δηλαδή να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά το ΣΥΖΑΡ, το TMS, προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση πρέπει να στηριχθεί παρετέρω. Θέλουμε να συνοδεύσουμε την κινητικότητα προς ε, τον αυτοματισμό της κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη νέες υπηρεσίες κινητικότητας. Και συγχρόνως το δίκτυό μας θα πρέπει να είναι περισσότερο ασφαλές και περισσότερο αντοχής απέναντι σε κλιματικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία, κάτι το οποίο δεν είναι παντεύκολο. Σχεδιάζουμε λοιπόν να προτείνουμε να καλύψουμε και τα συνολικά δίκτυα όπου αυτό γίνεται. Αυτό όμως θα το πετύχουμε μόνο με συλλογική προσπάθεια. Και έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο μου που είναι η συνέργεια, η συνεργασία μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακός κλάδος για τον αυτοματισμό στην κινητικότητα. Θα υπάρξουν δυνατότητες για τέτοια συνεργασία με ένα πλαίσιο όσο γίνεται πιο ανοιχτό στην συνέργεια, οπότε εκεί θα υπάρξει κατάλογος αλλά με αρκετή ευελιξία. Και το τρίτο μου σημείο έχει να κάνει με το κονδύλιο συνοχής. Μετά από τις πρώτες θετικές εμπειρίες, πρότεινε η Επιτροπή να μεταφέρει 11,2 δισεκατομμύρια από τη συνοχή στο συνδέοντας ε, την Ευρώπη βάσει των κανόνων. Βέβαια θα υπάρξει ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπως προβλέπετε. ενισχύοντας περισσότερο τις διασυνοριακές προσπάθειες. Τέλος, έρχομαι στο Invest EU και το μείγμα χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συγχώνευση των χρηματοδοτικών ε, μέσων που έχουμε τώρα σε ένα επενδυτικό. Ε, θα προβλέπετε κάτι για τις μεταφορές και θα συμπληρωθεί το συνδέοντας την Ευρώπη, εκεί όπου δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα. Θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα μίγματος χρηματοδοτικού με επιχορηγήσεις και άλλα μέσα ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, το νέο στοιχείο του συνδέοντας στην Ευρώπη, που είναι η στρατιωτική κινητικότητα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της νέας πρότασης που έχει γίνει για την άμυνα. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται προϋπολογισμός στο συνδέοντα στην Ευρώπη για να στηρίξει στρατιωτικές υποδομές ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα. Επινδύσεις λοιπόν που χρειάζονται για την κινητικότητα στον στρατιωτικό τομέα θα χρησιμοποιηθούν και για μη στρατιωτικό τομέα. Και το τελευταίο μου έχει να κάνει με την ενέργεια. Οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτούν χρηματοδότηση στις ε, υποδομές. Να μην χρησιμοποιούμε πια άνθρακα. Δίκτυα περισσότερο ψηφιοποιημένα και πιο ευφύ για να μπορεί να γίνει καλύτερα και η διαχείρισή τους. Κάποια δίκτυα μπορεί να τροποποιηθούν για συνθετικό αέριο ή για άλλες μορφές ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπώς, θα απαιτείται χρηματοδότηση και επενδύσεις. Εκεί κυρίως που οι υποδομές προβλέπουν και αυτό που λέμε externalities. Και το συνδέοντας στην Ευρώπη έχει να παίξει εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, χρειάζεται ένα φιλόδοξο κονδύλι και στήριξη για συνέργειες, όπως είπα και πριν. Μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακός κλάδος. Επιπλέον, πρέπει το συνδέοντας στην Ευρώπη να στηρίξει και άλλα επενδυτικά προγράμματα υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας. Συνεπώς, έχουμε ξεκινήσει για ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό συνδέοντας την Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να βασιστώ σε εσά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να προχωρήσουμε μαζί. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για 1,5 λεπτό ο κύριος Μαρινέσκου έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες τις οποίες μόλις μας δώσατε. Είναι σαφώς ότι οι υποδομές στον τομέα της ενέργειας και των τελεπικοινωνιών είναι η ουσία είναι κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούν ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών ή στον τομέα των αεναρίων μεταφορών και γι' αυτό ακριβώς θα μπορέσουμε να διασώσουμε τον μηχανισμό ακόμα και μετά από το 2021, 2021 αν και υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την αξιολόγηση των σημερινών τιμών, των τρεχουσών τιμών. Νομίζω πάντως ότι οι νέοι κανονισμοί θα τα διευκρινίσουν όλα αυτά. Να σας θυμίσω ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει 50 δις Αυτά που προτείνονται τώρα είναι λιγότερα από αυτά που ε, είχαν προταθεί το 2011 και ιδιαίτερα για τις μεταφορές. Για την ενέργεια έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, έχουν υπάρξει επίσης κάποιες βελτιώσεις και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μέχρι τις 6 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μία προσπάθεια για να αυξήσει τα διαθέσιμα χρήματα. Ευχαριστώ εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνάδελφος Σέντερ. Είναι σαφές ότι θα θέλαμε εμείς ε, να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και έτσι το σύνολο του Κοινοβουλίου να έχει μία κοινή θέση η οποία να οδηγήσει σε ισχυρές λύσεις για την επόμενη δεκαετία. Έχουμε σαφέστατες ελλείψεις στον τομέα των επενδύσεων σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και γι' αυτό ακριβώς οι προτάσεις αυτές μπορούν να είναι μια σημαντική βοήθεια για την επόμενη περίοδο. Οι προβλέψεις είναι σχετικά ρεαλιστικές. Υπάρχει μια μείωση βέβαια των προϋπολογισμών κατά 12 με 13% και αυτό είναι αναμενόμενο. Απαιτείται όμως να υπάρξουν συνέργειες κατεπίγουσες σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, τα λεγόμενα καθαρά αυτοκίνητα παράγονται πλέον και το θέμα είναι να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο. Και ζητάμε επίσης και ε, να υπάρξουν προσαρμογές στις χώρες των οποίων τα εθνικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στους συνολικούς στόχους. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος των συντηρητικών και ευρωπαίων μεταρρυθμιστών δίνω το λόγο στον κύριο Ζλοτόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πολύ που θεωρείται σημαντικό το πρόγραμμα Συνδέοντας στην Ευρώπη. Αυτό είναι θετικό για την πολιτική συνοχής. Μετά το 2020 θα τεθεί το θέμα των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών γιατί υπάρχουν διάδρομοι που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στον τομέα μέσω της συνέχισης των έργων και της συνέχισης της σύνδεσης των διαδρόμων αυτών. Αυτό θα προωθήσει την κινητικότητα, την αυτοματοποίηση διότι η πρωτοβουλία συνδέοντα την Ευρώπη περιλαμβάνει προγράμματα ε, και μηχανισμούς χρηματοδότησης που δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πέσουν θύματα της πολιτικής ε, λιτότητας. Περισσότερα χρήματα λοιπόν κύριε Επίτροπε. Τελίτσκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε αύριο. Σίγουρα θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι με τους συναδέρφους και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρω και εμείς στηρίζουμε τις δικές σας προσπάθειες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αρνητικά μηνύματα το συνδέοντα στην Ευρώπη είναι μια ιστορία επιτυχίας. Όλοι συμφωνούμε, αλλά πρέπει να δούμε πού πάνε τα κονδύλια και τότε διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περικοπέ. Και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι περισσότεροι εδώ, δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Τώρα για την αξιολόγηση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα αξιολογώντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, ώστε να μπορούμε να το δείξουμε στον κόσμο, στο κοινό, στους ανθρώπους. Το θέμα δεν είναι να του πούμε πόσα χρήματα δώσαμε, αλλά τι αποτελέσματα είχαμε. Τώρα, η περίπλοκη σχέση με το Horizon 2020 ή το EFSI, το επενδυτικό ε, σχέδιο Juncker. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε πως ή θα πετύχει ή θα το χάσουμε. Ή θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά ή θα πάνε περίπατο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ηλικιώτης, εκ μέρους της ε, ΚΟΕ, NGL. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν αξιοποιηθεί σωστά το πρόγραμμα συνδύοντας την Ευρώπη, μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών ενέργεια και μεταφορών που είναι ζωτική σημασία για του λαού τη ευρώπη. απαιτείται λοιπόν να πάψουν οι περικοπέ και να σταματήσει να διατίθεται μέρο του κονδυλίου στο ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων το οποίο αντί να προωθεί έργα δημοσίου συμφέροντο, επενδύει εκεί που συμφέρει στου ιδιώτες επενδυτέ. Το σημαντικότερο όμω είναι να μην χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό για την περαιτέρω στρατηγικοποίηση της Ένωσης μέσω της χρηματοδότησης υποδομών μεταφοράς για βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας όπως έχει εξαγγείλει η κομισιόν. στόχος πρέπει να είναι να προωθούνται έργα που έχει πραγματικά ανάγκη η κοινωνία τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς και στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα πληρούν όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες μια σημαντική προτεραιότητα είναι να προωθηθούν έργα για άρση της απομόνωσης στην οποία είναι καταδικασμένα ορισμένα κράτη και περιοχές στην ένωση. ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακαλώ. για Ο κύριος Φαντεκάμπ τώρα έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα το βράδυ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα, το λεγόμενο ΣΕΦ, Διευκόλυνση Συνδέοντα την Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για τις μεταφορές αλλά και για την ε, ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Το τελευταίο καιρό έχουμε αποδείξει ότι ένα από τα καλύτερα επενδυτικά προγράμματα, το πιο επιτυχημένο, είναι ακριβώς αυτό που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρόκειται εδώ πέρα για επιδοτήσεις, πρόκειται καθαρά για επένδυση στο μέλλον από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεπώς η σημερινή συζήτηση είναι προκειμένου να πείσουμε την Επίτροπο Μπούλτς να δώσει την τελευταία όθηση στο πρόγραμμα αυτό και όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μαρινέσκου να το διευρύνουμε όσο γίνεται. Πρόκειται πραγματικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει τον κόπο σήμερα έστω και τόσο αργά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο μηχανισμός Connecting Europe δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Όταν μιλάμε για προγράμματα υποδομών, ελείπουν οι επενδύσεις και είναι έτσι δύσκολος ο προγραμματισμός. Και γι' αυτό λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά έτσι ώστε να προωθηθούν τα TNT με σωστό τρόπο. Το εύση από μόνο του μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι πάντως στην παρούσα φάση απαιτείται να έχουμε δίκτυα τα οποία να διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη σύνδεση των περιφερειών μεταξύ τους ακόμα και των αποτέρων γεωγραφικά περιοχών και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκολύνει όχι μόνο τους νέους διαδρόμους αλλά το σύνολο του, ε, των διασυνδέσεων. Σαλίνη ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η πρόταση την οποία προτείνει ο συνάδελφος Μαρινέσκου είναι κάτι το οποίο έχει σαν βασικό στόχο την επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διασφάλιση της συνδεσιμότητας, την διασφάλιση της καινοτομίας. Πέραν α, της συγκέντρωσης των επενδύσεων στις κεντρικές υποδομές θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος και για επιμέρους δραστηριότητες όπως τα εναλλακτικά καύσιμα, η ψηφιοποίηση, και η μη χρήση ε, διοξιδίου του άνθρακα. Δεν δικαιολογούνται λοιπόν οι μειώσεις των ε, πόρων. Το θέμα δεν είναι μόνο η ποσότητα των πόρων, αλλά η τυπολογία του μηχανισμού που χρησιμοποιείται. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται με πολύ συγκεκριμένους στόχους και όχι όπως γίνεται σήμερα. E Ευχαριστώ. Ξεκινώ την διαδικασία Catch the Eye. Πέντε έχουν ζητήσει τον λόγο. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μίλαν Μόντ. Έχετε το λόγο, Πρόεδρε. Οι υποδομές των μεταφορών είναι βασικό χαρακτηριστικό της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Connecting Europe το δίδει θέμενη αξία η βελτίωση των υποδομών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την περιφερειακή συνοχή, την πρόσβαση στις εσωτερικές αγορές των περιφερειακών ε, ζωνών. Είναι κινητήρια δύναμη θα έλεγα ανάπτυξης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα δίκτυα μέχρι το 2030. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην συνδεσιμότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη των ε, παράκτιων περιοχών της Δυτικής Ευρώπης με μέτωπο στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι μελέτες που γίνονται θα πρέπει να τροποποιήσουν τον λεγόμενο Ατλαντικό διάδρομο που επηρεάζουν το βορειοδυτικό τμήμα της ε, Ιβυρικής Χερσονήσου έτσι μόνο το Connecting Europe θα σταθεί στο ύψος των προκλήσεων. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη μετά το 2020 είναι πράγματι σημαντικός. Όμως πρώτα απ' όλα απαιτεί κονδύλια και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση κονδυλίων. πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνδεσιμότητα και την καινοτομία. ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των χωρών και των περιοχών οι οποίες είναι απομονωμένες. αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ελλάδα η οποία είναι στο ακρότατο σημείο της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά επίσης και για τα νησιά τα νησιά του αιγαίου τα οποία έχουν κυριολεκτικά αποκοπεί στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο και να υπάρξει χρηματοδότηση των λειτουργικών ενεργειών και δράσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο μέσα από το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. ταυτόχρονα συμφωνώ με την έμφαση για νέες υποδομές ή εξυγχρονισμό των υποδομών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιλουάγκα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι για περιττές υποδομές. Και γιατί, γιατί μέχρι τώρα έχει δώσει ένα σωρό λεφτά για ορυκτά. Έπειτα, η τελευταία επένδυση θα είναι για την ηλεκτρική σύνδεση Ισπανίας και Γαλλίας. Η σύνδεση αυτή πήρε 578 εκατομμύρια. Συγχρόνως όμως έγιναν 6.000 ε, μηνύσεις κατά. Οργανώνεται κοινωνία λοιπόν κατά. Η διασύνδεση αυτή θα κοστίσει πολύ περισσότερα τελικά και ποιος θα τα πληρώσει ο κόσμος. Σύμφωνα με τους ρυθμιστές, πάντα αυξάνεται τελική τιμή κατά 3,5% τουλάχιστον. Έπειτα δεν ε, βοηθιέται καθόλου το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί τελικά με τα νέα αυτά δίκτυα περιορίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης ολικών πάρκων. Οπότε δεν νομίζω τελικά θα είναι θετικό όλο αυτό. Ευχαριστούμε. Νόβακοφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε τον προϋπολογισμό για να διαφημίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του μηχανισμού συνδέοντας στην Ευρώπη, διότι στους δρόμους της Ευρώπης περισσότερο πολιτική έχουμε παρά άσφαλτο και όλοι συμφωνούμε ότι η μεγαλύτερη αιτία ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων είναι τα μποτιλιαρίσματα και το καλύτερο μέσο για την επίλυση αυτού του προβλήματος ε, είναι ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μισό εκατομμύριο για την ολοκλήρωση του δικτύου και ακόμη δεν δίνουμε τον κατάλληλο προπολογισμό για την πρωτοβουλία συνδέοντας την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε. Συμφωνώ και διαπιστώνουμε τώρα ότι έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιπλέον εργαλεία και να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη, να τα οθήσουμε, να δώσουν τις δυνατότητες να ολοκληρώσουν τα δίκτυα των μεταφορών το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιμέντα Λόπες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Σε περιπτώσεις όπως αυτή για το συνδέοντας στην Ευρώπη, τα δίκτυα έχουν προσφέρει και δυνατότητες για εταιρική σχέση, για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος όμως τελικά αυξάνεται για τον κόσμο. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι είναι καλές. Θέλουμε να ξέρουμε τι προπολογισμό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου μάλιστα ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής δεν προσφέρονται σε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η οποία προσπαθεί να βελτιώσει το μέλλον ε, του πληθυσμού. Η Επίτροπος Μπούλκα έχει τώρα το λόγο. President, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή, η οποία δείχνει ε, τις θετικές πτυχές ε, του τωρινού ε, μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη και την ε, προθυμία να αυξήσουμε τον προπολογισμό και τι προτεραιότητε για μετά το 2020. Η περίοδο μετά το 2020 θα είναι κέρια σημασία ε, για να εξασφαλίσουμε ε, τα δίκτυα μέχρι το 2030. Πολλέ βελτιώσει του συνδέοντα στην Ευρώπη 2 θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων. Σημείωσα ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας για προτεραιότητες και για συνέργειες ε, σε έργα υποδομών. Θα ε, σχολιάσω κάποια από τα σχόλιά σας. Καταρχήν για τον προϋπολογισμό του συνδέοντας στην Ευρώπη. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει μια ε, φιλόδοξη πρόταση για το μέλλον του ΣΕΦ. Είναι, λίγα, είναι ένα από τα λίγα προγράμματα και φτάνει ε, στο 30,6 δισεκατομμύρια μέχρι ε, το 2030, δηλαδή περίπου 30% περισσότερο σε σχέση με την περίοδο 2014-2020. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνει τη διατήρηση των υφιστάμενων στοιχείων του στην Ευρώπη, αλλά και επιπλέον ενισχύεται με ένα νέο πυλώνα στρατιωτικής κινητικότητας, στις δύσκολες εποχές ε, που σχετίζονται με την απόσυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη ως ένα μέσον που προσθέτει επιπλέον αξία, προστιθέμενη αξία στην ε, ε, Ευρώπη. Όλα, να τονίσω εδώ ότι όλα τα χρήματα που δίδονται στην στρατιωτική κινητικότητα αφορούν τη δυτή χρήση. Μιλάμε για μη στρατιωτική χρήση, μη στρατιωτικό εξοπλισμό, για μη στρατιωτικού σκοπού ε, και για ενίσχυση τη στρατιωτική κινητικότητα. Όσον αφορά τι συνέργειες, μεταξύ μεταφορών ενέργειας και ψηφιακού τομέα. Όλα αυτά θα εφαρμοστούν με ε, κοινά προγράμματα που θα δώσουν τη δυνατότητα στον υψηλότερο βαθμό συγχρηματοδότησης για τον κάθε τομέα. Θα οριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για τις συνέργειες αυτές. να τονίσω άλλη μια φορά ότι η αρχή του ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να μην το χάσουμε θα παραμείνει στο συνδέοντα στην Ευρώπη γιατί είναι μία από τις βασικές αρχές που ε, οδήγησε στα υψηλά αποτελέσματα κατά τα πρώτα τρία έτη της ε, θητείας της Επιτροπής. Πάνω από 90% επιτευξη αποτελεσμάτων είχαμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τα έργα προτεραιότητας γιατί αναφέρθηκε σε ένα σχόλιο Ευρωβουλευτού. Πολλά κράτη-μέλη πρότειναν ε, νέα τμήματα, αλλά δεν μπορούσαμε όλα να τα ε, αναλάβουμε. Πολλά από αυτά θα ληφθούν υπόψη εφόσον ευθυγραμμίζονται με το παράρτημα του κανονισμού. Σας ευχαριστώ και πάλι. που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω την δομή της πρότασής μας, η οποία αναμένεται για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υποστήριξή σας. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε και προσβλέπω στις συζητήσεις μας κατά τους προσεχείς μήνες σε συντονισμό με τους συναδέλφους μου στον τομέα της ενέργειας και της ψηφιακής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έκλεισε η συζήτηση.